με τον εισηγητή και τους υπόλοιπους και όλους εισηγητές, νομίζω ότι πλέον βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Υπάρχουν βέβαια σημεία στα οποία πρέπει να γίνει περαιτέρω συζήτηση και νομίζω ότι ένα εξ αυτών, ένα πολύ σημαντικό σημείο, είναι το γεγονός ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και το ρόλο του Edward Snowden στην όλη διαδικασία. Και νομίζω ότι αυτό δεν έχει γίνει επαρκώς μέχρι τούδε και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξεύρουμε μία λύση και για την κατάστασή του. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει λόγο στο θέμα αυτό και επειδή δεν μπορέσαμε να τον ακούσουμε εδώ στη διαδικασία θα πρέπει να επιτρέψουμε και στους Ευρωπαίους πολίτες και στα Εθνικά Κοινοβούλια να βρουν μια λύση και να προσπαθήσουν να λάβουν όλες τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες και τις οποίες δεν θα λάβουμε βεβαίως όσο βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και πρέπει να παραμείνει στη Ρωσία και να βρίσκεται σε αυτό το, ε, το περίεργο καθιστός ε, και επειδή ακριβώς εμπλέκεται και η Ρωσία μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να διευκρινιστεί η κατάστασή του. Επίσης, να πω ότι πρέπει να γίνει έντονη έκκληση και προς τις κυβερνήσεις και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο Υπουργών για να υπάρξει εξονυχιστικός έλεγχος από πλευράς μας. Υπάρχει μια παρανόηση. Ε, μέχρι σήμερα το μόνο που κάναμε είναι να ε, δείχνουμε προς την ε, Ηνωμένε Πολιτείε γιατί δεν αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν τα ίδια προβλήματα και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ κυρία Ένστ. Σας ευχαριστώ. Πρώτα επιθυμώ και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή ο οποίος σε σύντομο χρονικό διάστημα μπόρεσε σε συνεργασία μαζί μας με μια απίστευτη ταχύτητα, επαναλαμβάνω, προσπάθησε και κατόρθωσε μέσω των ακροάσεων να δημιουργήσει μια βάση που ε, επέτρεψε και τις τέξεις εκθεσεώς του. Το ανθρωπίνος δυνατό μπόρεσε και το έκανε. Είμαστε το μόνο κοινοβούλιο που κάνει κάτι παρόμοιο που καταθέτει τέτοιο έγγραφο και αυτό οφείλω να το πω και απέναντι στις ε, χώρες μέλη, οι οποίες έχουν ωστόσο πολλά που θα έπρεπε να είχαν κάνει. μόνο λησμονούμε άλλωστε ότι οι μυστικές υπηρεσίες δρούν στις χώρες μέλη και έχουμε αφήσει και απ' τη βρετανική πλευρά. Και σε ό,τι αφορά την παραβίαση δικαίου Τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και αυτό ένα προβληματισμό στον οποίο πρέπει να εμβαθύνουμε και του επόμενου μήνε και όχι μόνο σε σχέση με την, του, την έκθεση πρέπει να τον αγάγουμε ω θέμα, να τον αγάγουμε σε θέμα. Εν τέλει το πρόβλημα είναι ποια θα πρέπει να είναι τα καθήκοντα των μυστικών υπηρεσιών και γιατί τις χρειαζόμαστε τις μυστικές υπηρεσίες. Εγώ δεν λέω τώρα εντελώς μπανάλ αν θα πρέπει να τις καταργήσουμε ή όχι, αλλά ποια θα πρέπει να τα καθήκοντά τους και ποια όχι. κατά πόσο η δράση τους επηρεάζει αρνητικά το κράτος δικαίου. Και αυτές οι εξουσίες τις οποίες έχουν από μόνες τους οικειοποιηθεί οι μυστικές υπηρεσίες. Όλα αυτά είναι κίνδυνος για τις ελευθερίες. Βέβαια σε, αυτή, σε αυτό τον προβληματισμό δεν μπορέσαμε να εμβαθύνουμε. Τέλος πάντων προσπαθούμε να βάλουμε στην έκθεση ό,τι μπορούμε. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία η έκθεση αυτή και από τις πλέον σημαντικές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ελπίζω να μπορέσουμε να εγκρίνουμε εν τέλει. Ποια είναι τα θέματα που για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Βέβαια, θα πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να υπάρξει απαγόρευση οποιονδήποτε μη ενδεδειγμένων ή περιττών συλλογών μαζικών δεδομένων. Έχουμε κάνει σχετικές συζητήσεις και στα πλαίσια του πακέτου για την προστασία των δεδομένων είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα αυτά. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εν τέλει και τι σημαίνει εθνική ασφάλεια. Πρέπει να καταφέρουμε τα επόμενα χρόνια να συζητήσουμε, να ορίσουμε την εθνική ασφάλεια. Τι ρόλο θα παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή θα λέμε μονίμως και διαρκώς «Α, δεν έχουμε εμείς καμία σχέση, είναι καθήκον των χωρών μελών». Δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλά τα πράγματα. Κάτι που δεν μου αρέσει και δεν έχει τόση σχέση με την ε, έκθεση όσο με τις συζητήσεις είναι όλη αυτή η φιλολογία γύρω από την εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών που πρέπει να αποκατασταθεί κτλ. Είπα ότι από την αρχή ότι για μένα αυτό είναι πρόβλημα. Εδώ οι δύο πόλοι είναι κυβερνήσεις και πολίτες. Πρέπει να το δει κανείς καθαρά αυτό. Οι πολίτες, οι πολίτες πρέπει να έχουν να μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στα συστήματα που τους διοικούν και βεβαίως και στις κυβερνήσεις. Αλλά όχι όλη αυτή η φλιαρία γύρω από την αιωνιότητα της πίστης φιλίας κατά τα λοιπά. Δεν μπορούμε να είμαστε υποτακτικοί των Ηνωμένων Πολιτειών. Εμείς τα απορρίπτουμε αυτά τα πράγματα. Και μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Βλέπω ότι υπάρχει το πρόβλημα αυτό, λιγότερο στην έκθεση. Κάποια, κάποιες επιπτώσεις, κάποιες συνέπειες πρέπει να υπάρξουν. Ναι, δεν θέλουμε safe harbor, τι είναι τα PNA και τα λοιπά, δηλαδή ανταλλαγέ δεδομένων επιβατών και τα λοιπά, ε, σχετικέ συμφωνίε, να τα αμφισβητήσουμε αυτά απέναντι στι ΗΠΑ. Τι άλλο έχουμε να πούμε εκτός από ωραία λόγια. Γι' αυτό είναι σημαντικό να δείξουμε καθαρά τι θέλουμε. Τώρα, η ασφάλεια των δεδομένων εντό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άλλο μέγα πρόβλημα αυτό. Και με υψηλό κόστο. Τα ακούσαμε αυτά. Να μπουν λοιπόν σχετικά κονδύλια στον προπολογισμό. Και τελευταία μου σκέψη, μακάρι να έχαμε και μια υποεπιτροπή στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προστασία δεδομένων. Αυτά για τον Σνόντεν τα είπε ο προηγούμενος. Ευχαριστώ. Τώρα θα μιλήσω από την ιδιότητά μου ως ε, εκπρόσωπος των φιλελευθέρων. Να ευχαριστήσω λοιπόν ε, τον εισηγητή, δεδομένου και του χρόνου, της χρονικής συγκυρίας των αποκαλύψεων και του πόσο διάστημα χρειάστηκε για να συνταχθεί η έκθεση, νομίζω ότι είναι προφανές ότι κάνουμε συστάσεις το επόμενο κοινοβούλιο, ώστε να ετοιμάσει αυτό με τη σειρά του ένα σχέδιο δράσης. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο μόνος φορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που διερευνά την όλη υπόθεση. Μόνο εμείς. Οι ίδιε οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν κάνει πολύ περισσότερα προκειμένου να διευκρινίσουν την κατάσταση από όσα έχει κάνει η Ευρώπη. Και επομένω, Νομίζω ότι αυτή η συνεχή σιωπή των κυβερνήσεων, το γεγονός ότι αρνούνται ε, να το συμπεριλάβουν ε, στο θεματολόγιο του Συμβουλίου ή σε συνεδριάσεις των ε, Υπουργών, θεωρώ ότι είναι σκανδαλώδες. Πολλό δε μάλλον, διότι είναι σαφές ότι ε, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι βλεγμένα στην υπόθεση. Είτε χρη, συνεργάζονται τα ίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε έχουν δικά τους συστήματα μαζικής παρακολούθησης. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να συνεχιστούν αυτά τα θέματα στην επόμενη θητεία, διότι αναμένουμε πολύ περισσότερες αποκαλύψεις. Η υπόθεση της Μπέλγακομ, για παράδειγμα, την οποία διερευνά ε, η δικαστική αρχή στο Βέλγιο. Και είμαι βέβαιη ότι θα μάθουμε πολύ περισσότερα στα επόμενα χρόνια για την υπόθεση. Όσον αφορά τώρα τις συστάσεις, κάποιες από αυτές κατά την άποψή μου είναι ζωτική σημασία. Καταρχάς θα πρέπει να αποκαταστήσουμε ή να ενισχύσουμε την νομική προστασία των Ευρωπαίων πολιτών. Δεύτερον, να ενισχύσουμε την εποπτεία των υπηρεσιών πληροφοριών σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τρίτον, και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό, να επενδύσουμε σε ασφάλεια δικτύων ε, πληροφορικής ε, την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής που διαθέτουμε. Τρι... Τέταρτον, πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι ιδίω οι πιο ευάλωτες ομάδες, ομάδες οι οποίες είναι πιο εκτεθισμένες και διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο κράτος δικαίου, πρέπει να προστατεύονται. Παραδείγματο χάρη δημοσιογράφοι, νομικοί, πολιτικοί, ε, δημόσια πρόσωπα εν γέννη, whistleblowers, πληροφοριοδότες, ακόμα και γιατρούς πέμπτη παρατήρηση για τις διεθνείς συμφωνίες. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να τις αναστείλουμε όλες αμέσως, διότι είναι μηδενικής αξίας. Και αν τα κράτη-μέλη τις θέλουν σώνη και καλά αυτές τις συμφωνίες, τότε πολύ σύντομα μπορούν ε, να μας δώσουν τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Και τέλος, δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις Ηνωμένε Πολιτείες, οι Ηνωμένε Πολιτείε κάνουν ό,τι κάνουν και οι υπόλοιποι. Απλώ έχουν καλύτερε δυνατότητε. Τα κράτη-μέλη το ίδιο κάνουν. Η Ρωσία το ίδιο κάνει. Ε, ξέρουμε τι γίνεται τις, ε, με τι μαζικέ ε, παρακολουθήσει, το, τη άτσι, τις ε, συλλογή δεδομένων αλλά και την αποθήκευση δεδομένων. Σήμερα ακούσαμε στα ειδήσει ότι ε, η Ρωσία παρισφρεί σε όλα τα συστήματα πληροφορικής. Η Κίνα είμαι σχεδόν βέβαιη ότι κάνει τα ίδια και άλλες χώρες. Ε, χώρες. Δεν χρειάζεται λοιπόν να επικεντρωθούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αρχή είναι αυτή η οποία μας ενδιαφέρει. Η κυρία Κορατσαμπίλ τώρα και έχω και άλλους τρεις ομιλητές. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον σκιώδη της Άλντε, με την σκιώδη της ότι πρέπει να βασιστούμε σε αρχές και να μην αναφερθούμε ιδιαίτερα σε κράτη. Και ενδιαφέρον μου προξένησε το γεγονός ότι αναφερθήκατε δικά στη Ρωσία, η οποία δεν ενέχεται σε όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες των πολιτών τι ανησυχίε του για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται και χρησιμοποιούνται δεδομένα. Και αυτό είναι μια σοβαρή συζήτηση την οποία πρέπει να την ε, διεξάγουμε, την, την διεξάγουμε ήδη και συγχαίρω τον κύριο Μωράης για το έργο του. Συμφωνώ ότι η μαζική παρακολούθηση δεν αφορά μόνο την εθνική ασφάλεια. Είναι φυσικά ζήτημα θεμελιωδών δικαιωμάτων και προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Θέλω να εκφράσω τις ε, ανησυχίε μου, τις οποίες προσπάθησα να ε, τονίσω και μέσω των τροπολογιών μου. Δεν θα πρέπει να συγχαίουμε την λειτουργία μιας επιτροπής διαρευνητική με μια δίκη, ούτε το Κοινοβούλιο είναι δικαστήριο. Θα πρέπει να είμαστε αυστηροί με τα κράτη-μέλη, με τις δραστηριότητες των κρατών μελών, αλλά δεν βρισκόμαστε εδώ για να απονείμουμε ποινές να καταδικάσουμε κάποιον. Γι' αυτό θεωρώ ότι οι διατυπώσει οι οποίες διαθέτουμε δεν είναι επικοδομητικές. Θα πρέπει να περιοριστούμε και να ακολουθήσουμε μάλλον το ρόλο που έχουμε ως θεσμικό όργανο ο οποίο βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Και να μην δημιουργήσουμε όργανα ή οποιασδήποτε διαδικασίε οι οποίε στην πραγματικότητα παραβιάζουν την αρχή της επικουρικότητας και δίνουν το μήνυμα στα κράτη-μέλη ότι συλλήβδην τους, ε, τα υποπτευόμαστε. Θα ήθελα λοιπόν να μου εξηγήσετε ποιος, ποια θα ήταν η προστιθέμενη αξία τη δημιουργία ενό τέτοιου οργάνου. Υπάρχουν τα εθνικά κοινοβούλια στα κράτη-μέλη, διαφορετικά κοινοβουλευτικά συστήματα και διαφορετικά συστήματα ελέγχου. Φυσικά και χρειάζεται ο δημοκρατικό έλεγχο, φυσικά χρειάζεται η λογοδοσία των εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών, αλλά δεν πιστεύω, μάλλον είμαι σίγουρη ότι ο χειρότερο τρόπο που θα μπορούσαμε να το κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε τέτοιου μηχανισμού ελέγχου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ προσωπικά σέβομαι τον τρόπο που έχουν επιλέξει τα κράτη-μέλη το καθένα να διεξάγει αυτόν τον έλεγχο. Εάν δεν συμφωνούμε με την κατάσταση σε κάποιο κράτος, μπορούμε να ζητήσουμε μεταρρυθμίσεις. Αλλά όχι να δημιουργήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα, ένα όργανο που δεν θα έχει καμία αξιοπιστία. Έχει σημασία η αξιοπιστία όταν αντιτιθέμεθα με τα κράτη-μέλη. Και θα ήθελα να σα φέρω το παράδειγμα τη Σουηδία μια και μιλάμε για ε, η νομοθεσία η σχετική για την προστασία της ιδιωτικής ζωής ε, υιοθετήθηκε μετά από πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση με ευρία πλειοψηφία το 2009 στο Σουηδικό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν πολλά, επίπεδα ελέγχου. Θα έλεγα μάλιστα ότι είναι υπόδειγμα για άλλους που θέλουν να βελτιώσουν το σύστημα λογοδοσίας τους. Οποιοςδήποτε μπορεί να το εξετάσει το μοντέλο το δικό μας το Σουηδικό είναι δημόσια διαθέσιμο. Ένας από τους υποψηφίους των πρασίνων προσεκλήθη στο Κοινοβούλιο για να μιλήσει. Και φυσικά χρησιμοποίησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να κάνει την προεκλογική του εκστρατεία και για να ε, επιτεθεί εναντίον της κυβέρνησης, όπως συνηθίζει η αντιπολίτευση. Και χρησιμοποιούμε την ε, ε, ομιλία του σαν να πρόκειται για μαρτυρία. Ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν πολιτικό ο οποίος απλώς επιτίθεται εναντίον της κυβέρνησης του, ως συνήθως και το χρησιμοποιούμε αυτό σαν να ήταν ε, αξιόπιστο αποδεικτικό υλικό. Αυτό δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε ε, αξιόπιστο αποδεικτικό υλικό, το θεωρώ σκανδαλώδες. Επίσης πρέπει να ξανασκεφτούμε με ποιον τρόπο προσκαλούμε άτομα να ε, εμφανιστούν ως μάρτυρες σε μια διαδικασία διαρευνητική όταν στην πραγματικότητα χρησιμοποιούν το βήμα για πολιτικούς σκοπούς. Λέμε ότι δεν θέλουμε να Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ευρωπαϊκέ εταιρείε για να βεβαιωθούμε για την ασφάλεια του συστήματο μα. Αλλά ο τρόπο αυτό, ο κατακαιρματισμό του ίντερνετ είναι πολύ ε, επικίνδυνος δρόμος γιατί υποβαθμίζει, υπονομεύει την ελευθερία στο ίντερνετ. Δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα της ε, ε, προστασία τη προσωπική ζωή στην πραγματικότητα υπονομεύοντα την ελευθερία του λόγου στο, στο, στο ίντερνετ. Δεν μπορούμε για παράδειγμα να αποκλείσουμε από τι ε, διαδικασίε προμηθειών, δημοσίων προμηθειών εταιρείε από τι ΗΠΑ, εάν αυτέ είναι ανταγωνιστικέ ή καλύτερε από τι ευρωπαϊκέ σύμφωνα με του κανόνε που εμεί θεσπίσαμε. Επίση, κυρία Πρόεδρε, δεν θα πρέπει να επιτιθέμεθα διακρίτως όταν έχουμε να κάνουμε με τις σχέσεις μας με τους συμμάχους. Δεν πρέπει να επιτιθέμεθα για παράδειγμα τη συμφωνίες για ανταλλαγές δεδομένων επιβατών της PNR εάν δεν έχουν παραβιαστεί οι όροι της συμφωνίας PNR. Πρέπει να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση, η συζήτηση για την ε, συμφωνία ομπρέλα για, την ελεύθερο, για το ελεύθερο εμπόριο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Ομπάμα, όπω και εσεί παραδεχτήκατε, έχει ξεκινήσει μια ε, διαδικασία μεταρρύθμισης του συστήματος ε, των υπηρεσιών πληροφοριών και πρέπει να αναμείνουμε τα αποτελέσματα. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω να συνεργαστούμε για να, με επικοδομητικό τρόπο για να προστατεύσουμε τελικά την ιδιωτική ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστούμε. Ο κ. Σπίρκερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ ευχαριστώ τον εισηγητή Μωράης για την δέσμευσή του, για την ενθουσιώδη του εργασία και για την ενδιαφέρουσα έκθεση. Συμφωνώ με τον Άξελ Φως που είπε ότι στις λεπτομέρειες η έκθεση χρειάζεται κάποιες βελτιώσεις. Και αυτό επιθυμώ, διότι λέει στο κάτω της γραφής στην ημερήσια διάταξη consideration of amendments. Ελπίζω ο εισηγητής να σχολιάσει έστω σύντομα τις τροπολογίες. Από πλευρά μου τώρα συγκεκριμένε παρατηρήσει για τι τροπολογίε. Μια πρώτη παρατήρηση που γνωρίζουμε όλοι και γνωρίζει και ο Σνόντεν ότι υπάρχουν κατασκοπικές δραστηριότητες, ότι οι ΗΠΑ λόγω των τεχνολογικών δυνατοτήτων τους έχουν χρησιμοποιήσει κάθε εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους. Αυτό δεν θα πρέπει όμως να μας αποτρέψει από του να σκεπτόμαστε, όπως είπε η Πρόεδρος, ότι δεν είναι μόναχα οι ΗΠΑ, είναι και άλλες δυνάμεις οι οποίες τα ίδια κάνουν ίσως χωρίς να τις αντιλαμβανόμαστε, ίσως μάλιστα και πολύ εντατικότερα από ότι είμαστε στη θέση να υποθέσουμε επί του παρόντος. Ας μην παραπλανηθούμε λοιπόν, ας έχουμε υπόψη μας ολόκληρη την εικόνα. Δεύτερο, Γνωρίζουμε ότι η αντικατασκοπία είναι εθνική υπόθεση. Το ίδιο ήταν πάντοτε και η αστυνομική ε, δραστηριότητα. Όμως η συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών έχει αποδείξει την αξία της στην αστυνομική συνεργασία και μέσα από αυτή τη συνεργασία ξεπίδησε η Ευρωπόλ ως ευρωπαϊκός θεσμός διότι διαπιστώσαμε ότι η συνεργασία αυτή αποδίδει. Και αυτό θέλω να το τονίσω λοιπόν. Και για την υποδομή γνωρίζουμε ότι επειδή ακριβώ δεν έχουμε επενδύσει, εξαρτώμεθα από την αμερικανική υποδομή στον τομέα της ε, τεχνολογίας της πληροφορικής. Αυτό ας το έχουμε υπόψη αν θέλουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα στο μέλλον. Για αυτό εγώ έχω στοχεύσει με τις τροπολογίες μου σε αυτή την κατεύθυνση. Πρώτα Να είναι σαφές ότι δεν είναι μοναχά οι ΗΠΑ που τα κάνουν αυτά. Δεύτερο, προτείνω να ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο όπως και με την αστυνομική συνεργασία. Δηλαδή να συνεργαστούν οι εθνικές υπηρεσίες. Όχι να δημιουργηθεί απαραίτητα αμέσως ένας ευρωπαϊκός οργανισμός, ίσως αυτό αν αποδείξει ότι είναι απαραίτητο να γίνει. Αλλά να υπάρξει πρώτα μια συνεργασία των εθνικών υπηρεσιών έτσι ώστε να προστατευθεί ο Ευρωπαίος πολίτης, η ευρωπαϊκή επιστήμη, η ευρωπαϊκή οικονομία απέναντι στην έξωθεν κατασκοπία. Αυτό θα πρέπει να είναι δυνατό και θα μας επιτρέψει να βάλουμε και μια τάξη και στις εθνικές υπηρεσίες, οι οποίες αντί να συνεργάζονται καμιά φορά ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Μπορούμε λοιπόν να φτιάξουμε εδώ ένα είδος ευρωπαϊκής αντικατασκοπίας, αλλά βεβαίως πολύ σχηδή και πολύ πτυχή χωρίς να γίνει καμιά αναθεώρηση συνθήκης για την ώρα. Και το τρίτο, όπως είπαν και άλλοι πριν από μένα, για την υποδομή. Να επενδύσουμε. Δεν θα έχουμε την απόλυτη ανεξαρτησία, κάτι τέτοιο βέβαια δεν είναι δυνατόν κιόλα στα πλαίσια αυτής της τεχνολογίας. Ωστόσο να έχουμε μεγαλύτερη αυτονομία για να μπορέσουμε να επιτύχουμε και υψηλότερη ασφάλεια. Ευχαριστώ κύριε Πέρκερ. Τελευταίος είναι ο κύριος Μιλντερ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή Νομίζω ότι έκανε μια πολύ καλή έκθεση, η οποία αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις ε, της Επιτροπής. Και εγώ κατέθεσα αρκετές τροπολογίες και η βασική ανησυχία μου, και νομίζω ότι σε αυτό λίγο πολύ συμφωνώ και με τους προλαλήσαντες, είναι ε, ότι επικρίνουμε πάρα πολύ τους Αμερικανούς, ε, όλα αυτά ναι με δικαιολογημένα, αλλά πρέπει να αναπτύξουμε δικές μας δυνατότητες. Πρέπει να έχουμε δικά μας ε, στοιχεία, να συλλέγουμε εμείς τις πληροφορίες που απαιτούνται για θέματα ασφαλείας ε, και τη μάχη κατά της τρομοκρατίας μόνοι μας και μετά να συντονιζόμαστε όσο το δυνατόν πιο στενά με τους Αμερικανούς. Αλλά πρέπει να τις δίνουμε εμείς τις πληροφορίες. Δεν ε, μπορούμε να τις δίνουμε εμείς συλλήβδιν στην άλλη πλευρά και να τις κάνουν ό,τι θέλουν. Εμείς θα πρέπει να τους δίνουμε τις πληροφορίες που απαιτούν και θα πρέπει να μας το ζητούν πρώτα. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θέλει να λάβει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να σχολιάσει. Έχω τρεις εδώ εκπροσώπους στον κατάλογο. Δεν θέλει η Κομισιόν να λάβει το λόγο. Η Προεδρία του Συμβουλίου. Δεν βλέπω διάθεση. Εντάξει λοιπόν, να περάσουμε στον κύριο Μωράες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέει ο κύριο Πέρκε. Είναι πολύ περίεργο, ε, μάλλον ασυνήθιστο ο τρόπο που έγινε η συζήτηση. Πράγματι, στην ε, ημερήσια διάταξη καταγράφεται ότι θα συζητήσουμε για τι τροπολογίε. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι ακριβώ αυτό. Συζητούμε για το σύνολο τη ε, εισήγηση στι συναντήσει με του κοιόδης πηγαίνουμε περισσότερο σε μια συζήτηση επί τη ουσία, επί των λεπτομεριών των τροπολογιών. Και φυσικά τι έχω λάβει υπόψη μου ε, ε, εδώ στην συνεδρίαση της Επιτροπής είναι ο χώρος και το βήμα θα έλεγα για να εκφράσει ο καθένας τα κύρια σημεία της άποψής του. Δεν θα μπορούσα να εξετάσω τις τροπολογίες μία-μία. Θα προσπαθήσω λοιπόν να απαντήσω στις παρατηρήσεις που έγιναν, ξεκινώντας από εκείνες του κ. Μάλτερ και του κ. Βος στην αρχή. Γνωρίζουμε πολύ καλά το ζήτημα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο τρόπος που δομήσαμε το έγγραφο ήταν για να αναδείξουμε ακριβώ αυτά τα ζητήματα του Safe Harbor, του, του ε, EU Cloud. του Ευρωπαϊκού Υπολογιστικού Νέφους. Όπως είπε και η Πρόεδρο, απευθυνόμαστε στην, στο κοινοβούλιο που θα προκύψει μετά τις εκλογές. Φυσικά τα μέλη έχουν υποβάλει τροπολογίες που αναφέρονται στο cloud προσωπικά. Και χαίρομαι που ορισμένες αυτές τι τροπολογίες έχουν πρωτότυπες ιδέες. Το συζητάμε στι συναντήσει με τους κοιόδης. Στην πρώτη συνάντηση, για να είμαι ειλικρινής, Συζητήσαμε κυρίως για τις διακρατικές ε, ανταλλαγές δεδομένων, διασυνοριακές μάλλον και τη συμφωνία TFTP. Θα προσπαθήσουμε να συζητήσω συζητήσουμε με τους συναδέλφους που έχουν προτείνει τροπολογίες για να δούμε τι θα γίνει με την κάθε μια από αυτές, πώς θα τις περιλάβουμε. Προσπαθώ να το κάνω έτσι, να, να, να, να ακολουθήσω αυτή την τακτική γιατί είναι πολύ δύσκολο να γίνει μια τέτοια συζήτηση εδώ με πλήρη σύνθεση της Επιτροπής. Με την άδειά σας λοιπόν, να απαντήσω σε ορισμένες από τις παρατηρήσεις που έγιναν. Κύριος Βόσου. ακολούθησε πιστά την γραμμή που εκφράζουν και οι τροπολογίες που έχει καταθέσει το ΕΛΚ. Κατά βάση η έκθεση αυτή είναι το αποτέλεσμα πολύ και συζήτηση συζήτησης μεταξύ των μελών του Κοινοβουλίου που επιδίωξαν να βρουν συμβασμούς, ε, συμβαστικές διατυπώσεις, να, να αναλύσουν ποια είναι τα σημαντικά θέματα που πρέπει να παραμείνουν και στις συμβαστικές ε, τροπολογίες. Αναφερόμαστε σε όλες τις ε, διεθνείς συμφάσεις, σε ζητήματα αρχής επίσης. Και όλοι οι σκιώδεις γνωρίζουν πολύ καλά ότι πρόκειται για μια έκθεση ε, μιας διερευνητικής επιτροπής. Άρα δίνει και μια εικόνα, ε, μια, ένα αφήγημα στους Ευρωπαίους πολίτες, εξηγεί τι συνέβη. Την άποψή μας για το πώς έχουν τα γεγονότα. Γι' αυτό έχουμε καλέσει και τους ε, μάρτυρες και θέτουμε ζητήματα αρχής, θέτουμε τεχνολογικά ζητήματα και προσπαθούμε στις συναντήσεις ε, με τους σκιώδεις να καταλήγουμε σε σωστές συμβαστικές διατυπώσεις. Και αναφέρεται και το EU Cloud, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Νέφος, στις ε, συζητήσεις αυτές. Εδώ έχουν διαφορετικές θέσεις οι πολιτικές ομάδες. Ο, Γιάννης μίλησε για τον Σνόουντεν. Υπάρχουν και σχετικές τροπολογίες. Και εγώ το θεωρώ σημαντικό. πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποιε απόψει, ποια, ποια, θέματα θέτει κάθε πολιτική ομάδα και πώ τελικά καταλήγουμε σε αυτέ τις ε, συμβαστικέ διατυπώσει. Προσπαθώ να το κάνω αυτό όσο το δυνατόν πιο διεξοδικά και όσο το δυνατόν, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια. Με αυτά τα θέματα οφείλουμε να μιλάμε ανοιχτά. Είμαι σίγουρος λοιπόν οι επόμενες συναντήσεις των σκιωδών θα είναι πολύ εργόδης. Αλλά τι προσπαθώ να πω. Προσπαθώ να πω ότι χρειάζεται διαφάνεια. Πρόκειται για ένα ευαίσθητο πολιτικό θέμα για το Κοινοβούλιο και γενικότερα. Και το έθιξαν και ορισμένοι συνάδελφοι. Κανένα άλλο εθνικό κοινοβούλιο δεν ανέλαβε παρόμοια πρωτοβουλία. Κανένα άλλο εθνικό κοινοβούλιο, για παράδειγμα, δεν αναφέρθηκε σε όλη αυτή τη σειρά ζητημάτων που και τεχνολογικών και ζητημάτων εποπτεία, θεσμικών κτλ. Γι' αυτό ε, λοιπόν η πρόεδρος της τεχνολογίας μας έχει θέσει τέτοια επιτακτικά θέματα. κονίλια. Και εσείς αναφερθήκατε σε ορισμένα κρίσιμα θέματα. Εσείς αναφερθήκατε κυρίως στο μέλλον και πώς θα θωρακιστούμε καλύτερα στο μέλλον, πώς θα δημιουργήσουμε ένα σχέδιο δράσης που θα μας προστατεύει στο μέλλον. Και πάλι το σημαντικό εδώ είναι να δημιουργηθεί αυτό το σχέδιο δράσης και αυτός ο μηχανισμός που θα διαρκέσει, που θα παραμείνει. Αναφερθήκατε εσείς επίσης, στην στο... ρωτήσατε μάλλον ποια είναι η προσδεθέμενη. Παρεμβαίνει. Εγώ δεν ρώτησα για την προστιθέμενη αξία τη έκθεση. Εγώ ρώτησα ποια θα ήταν η προστιθέμενη αξία του να δημιουργηθεί ένα μηχανισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πολύ διαφορετικό, έτσι. απάντηση του κ. Μωράε. Θα υπάρχει εμπλοκή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Γι' αυτό συζητάμε. Η πρόεδρο, καλύτερα να μην μπαίνουμε σε τόσο πολλέ λεπτομέρειε. Κ. Μωράε, ναι, πράγματι. Οι τελευταίοι ομιλητέ, νομίζω, έχουν υποβάλει τροπολογίες που τις καλωσορίζω. Έχει υπάρξει πολλή σκέψη επ' αυτόν. Αυτό που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι ότι θα προσπαθήσω να τις συμβιβάσω με όσο το δυνατόν ε, διαφανέστερο τρόπο. Υπάρχουν κάποιες ε, ε, τροπολογίες οι μπαίνουν πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και θα πρέπει να είναι σαφές ε, πώς τελικά θα τις αντιμετωπίσουμε, τι θα κάνουμε με αυτές. Να ευχαριστήσω πάντως τους, τη, τη γραμματεία, το προσωπικό που έχει αναλάβει όλο αυτό το τιτάνιο έργο από την γραφειοκρατική πλευρά είναι σημαντικό γιατί εδώ πρόκειται για διερεύνηση της κατάστασης και να ευχαριστήσω λοιπόν τον προσωπικό και τους κοιόδης που έχουν αφιερώσει τόσο χρόνο στις συναντήσεις. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε. Είμαι βέβαιη ότι όλοι συμφωνούμε ε, με τα συγχαρητήρια που δώσατε στο προσωπικό και στη γραμματεία. Πράγματι γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο να βρίσκει κανείς συμβιβαστικές λύσεις όταν έχουν υποβληθεί τόσες πολλές τροπολογίες. Σίγουρα δεν γίνεται όταν η Επιτροπή ε, συνεδριάζει σε σώμα. Αλλά όπως είπατε κι εσείς, οι συναντήσεις των σχεδόν θα πρέπει να γίνονται με όσο το δυνατόν διαφανέστερο ε, ανοιχτό τρόπο. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ. Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσια διάταξης. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ομάδα δράσης για την Μεσόγειο. Ο κύριος Μούσολ ήταν ο... Μάσελ, είναι, είναι ο υπεύθυνο ορμόδιο ε, για αυτό το ζήτημα από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα. Επομένω, θα αναγκαστώ για τέταρτη φορά να διακόψω τη σημερινή μα συνεδρίαση για 10 λεπτά και θα ε, ξαναξεκινήσουμε στι 3. Colleagues. Σας παρακαλώ, καθίστε. Έχει έρθει ο κύριος Μούσελ και γι' αυτό να καθίσετε πάλι και όποιοι επιθυμούν να συζητήσουν παρακαλώ εκτός. Ωραία λοιπόν. Μετά από, τον, την αυτική τραγωδία στα νυχτά της Λαμπεντούσα τον Οκτώβριο του 2013 όπου πνίγηκαν παραπάνω από 360 άνθρωποι το Συμβούλιο αποφάσισε να φτιάξει μια ειδική ομάδα για τη Μεσόγειο με εντολή να εντοπίσει δράσεις κατά προτεραιότητα για πιο αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών πολιτικών και εργαλείων με σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 12 του 2013 που υπευλήθη για συζήτηση στο Συμβούλιο Τζάι στις 5 και 6 12 του 2013 και συζητήθηκε επίσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 19 και 20 12 του 2013. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγραψε επισήμως στην Επίτροπο Μάλμστρομ για να εκφράσει την λύπη του για την καθυστερημένη και ατελή διαβίβαση των πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις συναντήσεις της Task Force. Και στην βάση της συμφωνίας μεταξύ Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής ιδίω για συναντήσεις εθνικών εμπειρογνωμόνων όπου στο σημείο 2 του παρατήματος 1 λέει ότι η Επιτροπή αναλαμβάνει τη δέσμευση να διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο τα σχετικά έγγραφα καθώς και τις ημερήσιες διατάξεις στο mailbox του Κοινοβουλίου ταυτόχρονα με τη στιγμή που τη στέλνει στους εθνικούς εμπειρογνώμονες. Είμαι βεβαία ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φροντίσει ότι στο, ώστε στο μέλλον οι πληροφορίες αυτές να διαβιβάζονται σύμφωνα με την Συμφωνία Πλαίσιο. Έχοντας πει όλα αυτά, καλωσορίζω τώρα τον κύριο Μούσελ, Διευθυντή Μεταναστεύσεως και Ασύλου στην Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών, που θα ε, εξηγήσει τα σχετικά. Κύριε Μούσελ, έχετε το λόγο και νομίζω ότι διαθέτεται και διαφάνειες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και πρώτα να αντιδράσω στα όσα είπατε για την διαβίβαση των εγγράφων και μετά θα έρθω στο ουσιώδες περιεχόμενο. Η Task Force δεν θεωρήθηκε ως ομάδα εμπειρογνωμόνων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συναπαρτίζεται από 28 χώρες μέλη, συνδεδεμένες χώρες και 5 οργανισμούς σε υψηλό επίπεδο για να συζητήσει θέματα μετά τα συμβάντα της Λαμπεντούσα. Ήταν λοιπόν ένα ειδικό όργανο το οποίο δεν έχει προηγούμενο στα ιστορικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι εκτός πλαισίου συνθήκης. Αυτό λοιπόν που κάναμε είναι ότι προσπαθήσαμε να το ξαναφέρουμε μέσα στο πλαίσιο των επιτροπών. Εγώ ήμουν επικεφαλής της Task Force, μπόρεσα να πείσω τα μέλη της Task Force να συντάξουμε ανακοινοθέν από την Επιτροπή για να επανέλθει το θέμα μέσα στο θεσμικό πλαίσιο και αυτό που κάναμε ήταν μια ανακοίνωση για το έργο της Task Force που εμφανίζεται τώρα και ενώπιον, δηλαδή που στέλνει πλέον τα έγγραφά της και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Τώρα που έχει λήξει η εργασία της Task Force, έχει ολοκληρώσει το έργο της, έχει έλθει πλέον η ώρα του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου να εξετάσουν τις ε, διάφορες ε, δράσεις. Αυτή ήταν η θέση μας. Βέβαια θα μπορούσαμε να είχαμε ενημερώσει καλύτερα το Κοινοβούλιο και εκφράζω τη λύπη μου που δεν ήταν αρκετά σαφές αυτό πριν από τη σημερινή συνεδρίαση η πρόεδρος Ιντφέλτ, για να κατανοήσω καλά αυτά που λέτε, οι συναντήσει που ανέφερα έγιναν όχι στην βάση του ανακοινοθέντος της Κομισιόν και λάβαμε το έγγραφο ταυτόχρονα με το Συμβούλιο. Αυτό μου λέτε. Ναι, η ανακοίνωση της Επιτροπής διαβιβάστηκε ταυτόχρονα στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Το έργο της Task Force είχε ολοκληρωθεί ήδη. Και το ανακοινοθέν εξήχθη από αυτό το έργο της Task Force. Εσείς ζητάτε να σας είχαμε κοινοποιήσει το έργο της Task Force στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά όπως είπα ήταν ειδικό όργανο, εμείς ρωτήσαμε την νομική μας υπηρεσία, μπορεί βέβαια κανείς να έχει και διαφορετική άποψη, διαφορετικές απόψεις ίσως των νομικών υπηρεσιών, αλλά αυτή ήταν η θέση που μας υποβλήθηκε τότε. Αλλά ίσως είναι καλύτερα να προχωρήσουμε στην ουσία που ίσως είναι και πιο σημαντική από τη διαδικασία ναι, όχι, οι διαδικασίες όμως μετρούν, διότι οι διαδικασίες είναι αναπόσπαστο μέρος της, διαδικασίας, της ε, δημοκρατίας. Λάβαμε βέβαια 15 μέρες αργότερα και την ημερήσια διάταξη και όλα τα σχετικά. Αλλά λέτε τα ίδια και, όταν, ε, και θα λέμε τα ίδια όταν δημιουργούνται όργανα εκτός των ε, πλαισίων των συνθήκων. Ενώ εμεί προτιμούμε την κοινοτική μέθοδο, όπω γνωρίζετε. Μάλιστα, α προχωρήσουμε στι διαφάνειέ σα. Ευχαριστώ. Για την ίδια την ε, Task Force δημιουργήθηκε μετά από την τραγωδία της Λαμπεντούσα που ήταν ε, ένα, κάτι που μας αφύπνισε. Έχω λίγες διαφάνειες που μπορώ να σας δώσω βλέπετε και την λίστα των γεγονότων 360 άτομα που ε, πέθαναν στις 3 Οκτωβρίου, μετά από λίγο έγινε το Συμβούλιο Τζάι και ε, εκεί αποφασίστηκε να ιδρυθεί η Task Force, η οποία έλαβε υπόψη και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα δείτε και στην ανακοίνωσή μας ότι παραπέμπουμε και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Task Force λοιπόν ως στόχο είχε να εξετάσει βραχυπρόθεσμες δράσεις, βραχυπρόθεσμες, όχι μακροπρόθεσμες λύσεις. Εντόπισε λοιπόν πέντε είδη δράσεων. Πρώτη, συνεργασία με τρίτες χώρες. Δεύτερο, περιφερειακή πρόταση, resettlement. τρίτη, ο αγώνας κατά των δουλεμπόρων. Τέταρτο, η εποπτεία των συνόρων και η τελευταία αλληλεγγύη προς τις χώρες που βρίσκονται ας πούμε στην πρώτη γραμμή του πυρός, έτσι να το πω έτσι. Τώρα, για τη συνεργασία. Το νέο στοιχείο εδώ είναι ότι για πρώτη φορά οι Υπουργοί Εξωτερικών και η Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων λαμβάνουν υπόψη σοβαρά τα θέματα της μετανάστευσης, διότι δεν ήταν υψηλά ε, στις προτεραιότητες και τώρα μπαίνουν πολύ υψηλά στις προτεραιότητες Εργαζόμαστε λοιπόν, συνεργαζόμαστε με τρίτες χώρες, με την Ισία. Προχωρούμε σε συμφωνίες συνεργασίας με ένα αριθμό τρίτων χωρών. Αυτό που χρειάζεται ωστόσο είναι σαφής, συγκεκριμένη δράση επιτόπου. Παράδειγμα, πολλοί φεύγουν από την ε, Σαχάρα, περνάνε μέσω Λιβύης. Δεν υπάρχουν αρκετά σκάφη διότι όταν τα βρίσκουν τα σκάφη τα κατάσχουν οι border guards. Υπάρχει λοιπόν τώρα ένα εμπόριο μεταξύ την Ισίας και Λιβύης σκαφών. Είναι πολύ δύσκολο για την ώρα να έρθουμε σε επαφή και να συνεργαστούμε με τις λιβικές αρχές. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με τις τινησιακές αρχές για να πάψει το εμπόριο μεταξύ Τινησίας και Λιβύης για σκάφη. Να λοιπόν μια συγκεκριμένη δράση για να σας ε, εικονογραφήσω το τι πρέπει να κάνουμε επιτόπου. Το ίδιο εκστρατείες ενημέρωσης, πληροφόρησης από τα κύρια στοιχεία που τόνισε η Task Force να ενημερωθούν οι μετανάστες στις χώρες προελευσής τους, στις χώρες διαβασής τους για τους κινδύνους που αναλαμβάνουν φτάνοντας παράνομα στην Ευρώπη ή προσπαθώντας να φτάσουν παράνομα στην Ευρώπη. Πολλοί χρεώνονται για να φύγουν από εκεί, πληρώνουν οι, οικο, οικογένειες, βιάζονται οι γυναίκες και ούτω καθεξής. Πρέπει λοιπόν να ενημερωθούν τα πρόσωπα αυτά για τους κινδύνους και βέβαια να υπάρξουν και περισσότερα νομικά κανάλια για να αντιληφθούν ότι ε, να πληροφορηθούν για τους κινδύνους της παράνομης αυτής μετανάστευσης. Τώρα, χρειάζεται επίσης να ενισχύσουμε τα περιφερειακά προγράμματα προστασίας. Στην Βόρεια Αφρική και στην ε, γειτονία εκεί, να αναπτύξουμε επίσης περισσότερες πολιτικές επανεγκατάστασης, resettlement. Η Κομισιόν έχει ζητήσει κατ' επανάληψη από τις χώρες μέλη να αυξήσουν τα ποσοστά, τις ποσοστώσεις resettlement. Το πιο δύσκολο βέβαια θέμα της Task Force, διότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη διάθεση από τις χώρες μέλη να αυξήσουν τις νόμιμες οδούς, τους νόμιμους διάβλους για την έλευση στην Ευρώπη. Όταν μιλούμε για νόμιμη μετανάστευση, εποχικούς εργαζόμενους, σπουδαστές κλπ. Αυτά, εκεί υπάρχουν συγκεκριμένα νομικά όργανα, νομικά κείμενα που μπορούν να επιτρέψουν. Μιλούμε τώρα και για αυτούς που ζητούν άσυλο και επίσης για ανθρωπιστικές ε, προξενικές θεωρήσεις κλπ. που είναι επιλογές που μπορούν να αυξήσουν τις δυνατότητες νόμιμης μετανάστευσης. Και αυτά βεβαίως πρέπει να γίνουν και αντικείμενα μελετών. Επίσης, ο αγώνας κατά του οργανωμένου εγκλήματος των δουλευόρων εδώ ζητεί η Task Force από την Ευρωπόλ να προχωρήσει σε συγκεκριμένες δράσεις σε συνεργασία με, την Ευρωπαϊκή, με τις χώρες μέλη για να διαλυθούν τα δίκτυα. Πολύ δύσκολο βέβαια διότι τα δίκτυα αυτά οργανώνονται σε τρίτες χώρες. Επομένως η δική μας δυνατότητα παρέμβαση είναι περιορισμένη. Πρέπει όμως να συνεργαστούμε ιδίω με χώρες διάβασης όπως την Τινησία, το Μαρόκο, τη Λιβύη, την Αίγυπτο, την Τουρκία για να μπορέσουμε έτσι να αγωνιστούμε κατά των ε, ε, δουλεμπόρων. Η Κομισιόν επίσης αναθεωρεί την υφιστάμενη νομοθεσία, την επαρεξετάζει δηλαδή για να δει αν είναι αρκετά ενημερωμένη, αρκετά επίκαιρη και αν ίσως πρέπει να αναλυθούν κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Εν τέλει, η εποπτεία των συνόρων, επίσης κέριο θέμα, η επιχείρηση Mare Nostrum, η οποία ήδη έχει βελτιώσει σημαντικά την κατάσταση γύρω από την Ιταλία. Τα σκάφη δεν φτάνουν πλέον στην Λαμπεντούσα, στέλνονται στην ε, Σικελία και στον κύριο κορμό της Ιταλίας και έτσι έχουν σωθεί πολλές ζωές. Και υπάρχουν και επιχειρήσεις Frontex που συνεχίζονται. Έχουμε ενισχύσει τον προϋπολογισμό της Frontex κατά 7,9 εκατομμύρια ευρώ μόλις τον Οκτώβριο και προσπαθούμε να βελτιώσουμε και την εικόνα της κατάστασης στην περιοχή για να μπορούμε να εντοπίζουμε τα σκάφη που χρειάζονται διάσωση. Κάνουμε πρόοδο επίσης και με τον κανονισμό ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια μέσα τα χρονικά πλαίσια της ελληνικής προεδρίας για την λειτουργία της Frontex. Οι πιθανότητες είναι αρκετά καλές, να είναι ξεκάθαρο δηλαδή ποιος κάνει τι στην περίπτωση αποβίβασης ε, προσώπων. Επίσης, τέλος, αναλαμβάνουμε πολλές δραστηριότητες, το 5 λέω τώρα, για την αλληλεγγύη και στήριξη των χωρών μελών. Έχουμε κινητοποιήσει έκτακτα κονδύλια για την Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Ιταλία τις χώρες που είναι στην πρώτη γραμμή δηλαδή, βελτιώνοντας έτσι τις δυνατότητές τους να υποδεχθούν πρόσφυγες. Όπως ξέρετε, 10.000 άνθρωποι φτάνουν στην Βουλγαρία, από, έφτασαν από τον Σεπτέμβρη μέχρι τον Δεκέμβρη, μαζική ροή λοιπόν, για να μπορέσει η χώρα αυτή να αντιμετωπίσει τις ροές αυτές ορθά. Σημαντική πίεση σημειώνεται και στην Ιταλία, έρχονται οι βάρκες ακόμα τώρα τον χειμώνα και εκεί έχουμε προσφέρει έκτακτη ε, βοήθεια στη χώρα αυτή. Θέλω να τονίσω ακόμη ότι αλληλεγγύη σημαίνει και ευθύνη. Λαμβάνεται λοιπόν ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις χώρες μέλη, εφόσον η συγκεκριμένη χώρα που δέχεται την ε, βοήθεια εφαρμόζει το κοινοτικό και εκτιμένο πλήρως. Το επόμενο βήμα ή τα επόμενα βήματα εν συμπεράσματι θα πρέπει να είναι η φάση της εφαρμογής όπου θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο επιχειρησιακοί επιτόπου. Η Κομισιόν δουλεύει με τις χώρες μέλη, με τους αρμόδιους οργανισμούς για να εξασφαλίσουν ότι η ανακοίνωση δεν θα παραμείνει στα χαρτιά αλλά θα αποτελέσει ένα πραγματικό επιχειρησιακό σχεδιασμό για την βελτίωση της κατάστασης και θα επανέλθουμε να υποβάλουμε τα σχετικά στο Συμβούλιο του Ιουνίου για την εφαρμογή της ανακοίνωσης. Πάμε και στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών μάλλον το Μάρτιο και τον Ιούνιο για να ενημερώσουμε σχετικά με τα βήματα που έχουμε κάνει μετά από την έγκριση της ανακοίνωσης. Και βέβαια πολύ ευχαρίστως θα ακούσουμε τις απόψεις σας και είμαστε και στη διάθεσή σας να επανέλθουμε ανα πάσα στιγμή για να σας ενημερώσουμε για το πού βρίσκεται η εφαρμογή των προτάσεων της Task Force. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Πριν δώσω το λόγο στην Προεδρία του Συμβουλίου, νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να μας ενημερώνετε τακτικά για την κατάσταση της εφαρμογής, διότι πλέον γνωρίζουμε ποιοι είναι οι στόχοι, ποιο είναι το σχέδιο, αλλά νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλό να παρακολουθούμε και την πρακτική εφαρμογή επιτόπου. Ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε να, ξα... να σας ζητήσουμε να έρθετε και πάλι σε ένα μήνα περίπου για να μας πείτε πού βρισκόμαστε με την έκθεση πρόοδου. Η Ελληνική Προεδρία θέλει να σχολιάσει. Ο κύριος ή ο κύριος Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου, εφόσον μου δίνετε δυνατότητα να μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα και ευχαριστώ πολύ για αυτό το Κοινοβούλιο. Ε, η Προεδρία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ε, άμεση εφαρμογή ε, των δράσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής και προτίθεται να επιβλέπει αυτή την εφαρμογή των δράσεων στα διάφορα όργανα του Συμβουλίου. Ε, στο πλαίσιο των δράσεων, για παράδειγμα, ε, περιλαμβάνεται και η ολοκλήρωση του κανονισμού για τη θέσπιση κανόνων διεξαγωγής κοινών επιχειρήσεων του Frontex στα θαλάσσια σύνορα και χαιρόμαστε που με τη βοήθεια και του Κοινοβουλίου προχωράμε και θα είμαστε ίσως σε θέση να το ολοκληρώσουμε ε, πριν από τις Ευρωεξτό. <laughs> Πολύ σύντομο ήταν αυτό. σα ευχαριστούμε. Έχει ζητήσει ένα συνάδελφος το λόγο. Ο κύριο Μιλτερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω ένα ερώτημα προ την Επιτροπή. Εάν κατάλαβα καλά, πρόκειται να υπάρξει διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας ε, μεταξύ μάλλον με τις χώρες που βρίσκονται στα σύνορα, στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, κυρίως τις μεσογειακές. Ο κανονισμός ίσως δίνει τη δυνατότητα να αποσπαστούν άτομα με συγκεκριμένη αρμοδιότητα στις πρεσβείες, στις αποστολές μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στις χώρες αυτές, με την αρμοδιότητα να αναφέρουν σε ζητήματα σχετικά με τις πρόσφυγες. Θα αξιοποιήσει η Επιτροπή αυτή ε, τη δυνατότητα που της δίνει ο κανονισμός. Δεύτερο ερώτημα, η Ιταλία. Ήταν από τις πρώτες χώρες που συμμετείχε στο πιλωτικό πρόγραμμα Eurosur. Ήταν μια χώρα η οποία δημιούργησε από πολύ νωρί ένα ε, κέντρο εθνικού συντονισμού. Παρ' όλα αυτά, η τραγωδία της Λαμπετούσα δεν αποφεύχθηκε. Πώς γίνεται, πώς μπορείτε να μου εξηγήσετε ότι η ίδια χώρα είναι εκείνη που ήταν η πρώτη που συμμετείχε στην Γιουροσούρα ε, αλλά παρ' όλα αυτά δεν αποφεύχθηκε η τραγωδία. Ωραία. εκτό και αν θέλει κάποιο άλλο μέλος να λάβει το λόγο, θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις. Ναι, σας ευχαριστώ. Όσον αφορά τον αξιωματικό σύνδεσμο, θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν να συστήσουμε δίκτυα αξιωματικών συνδέσμων σε τρίτες χώρες. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ καλή πρακτική και αν τα κράτη-μέλη ε, μπορούν να έχουν διαθέσιμους πόρους εκεί, τότε ε, θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε με την εξουσιοδότησή μας και νομίζω ε, ότι είναι πολύ καλή πρακτική. Στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου έχουμε αξιωματικούς συνδέσμους, για παράδειγμα, και μπορούμε να ε, δημιουργήσουμε συνέργειε επιτόπου. Όσον αφορά το ερώτημά σας για τη Eurosur και το γεγονό ότι η Ιταλία ήταν η πρώτη, ε, δεν κατάλαβα ακριβώς τι μήνυμα θέλετε να περάσετε. Ζητώ συγγνώμη. Νομίζω ότι ήταν θετικό το γεγονός ότι κινητοποιήθηκε η Ιταλία για το Eurosur και ε, ακολουθούν και άλλα κρατημέλη ε, και όλοι έχουν δεχτεί να συμμετέχουν. Ε, για μένα είναι θετικό το γεγονός ότι έκανε το πρώτο βήμα η Ιταλία. Ίσως δεν αντιλήφθηκα όμως ακριβώς το νόημα της ερώτησής σας. Δεν ικανοποιηθήκατε κύριε Μούλτερ. Ναι, για να διευκρινίσω. Αυτό που εννοούσα είναι ότι η Ιταλία ήταν η πρώτη η οποία συνεργάστηκε στο Eurosur και θα μπορούσαν να είχαν ειδοποιήσει και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη για βοήθεια και δεν έγινε κάτι τέτοιο. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι γιατί αφού το Eurosur υποτίθεται ότι βελτιώνει την επικοινωνία μεταξύ των κρατών μελών και σε αυτή την περίπτωση εγώ δεν είδα και καμία επικοινωνία. Κομισιόν. Well, so Αναφέρεστε στο συγκεκριμένο γεγονός, λοιπόν, στη Λαμπεντούζα τότε. Ναι, δεν αντιλήφθηκα την ερώτησή σας. Υπάρχει δικαστική έρευνα εν εξελίξη για το κατά πόσον διαπράχθησαν σφάλματα από τις Ιταλικές αρχές και από τους συνοριοφύλακες ε, στην περίπτωση αυτή. Δεν θα ήθελα εγώ να παρέμβω ε, στη δικαστική έρευνα, διότι όπως σας είπα είναι εν εξελίξη και ε, δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να είχαν ε, λάβει στήριξη από κάποιον άλλον τότε. Ε, αυτά τα πράγματα όταν φτάνουν πολύ κοντά στις ακτές της Λαμπεντούζα προχωρούν πάρα πολύ γρήγορα. Ίσως να μπορούσαν να είχαν κινητοποιήσει κάποιους άλλους για βοήθεια, αλλά δεν γνωρίζω. Αυτό επαφίεται στο δικαστή και αυτό θα ε, αποφανθεί για το κατά πόσον υπήρξε κάποιο σφάλμα. Ωραία, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε με αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστούμε τον κύριο Μούσελ και ελπίζω να μπορέσουμε να σας καλωσορίσουμε και πάλι εδώ στην Επιτροπή για να μας κάνετε μια έκθεση πρόοδου. Okay. Um, Ωραία. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Η έκθεσή μου για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα. Υποτίθεται ότι είναι ετήσια έκθεση, αλλά είναι για το διάστημα από το 2011 έως το 2013, επομένως είναι διετής. Είναι η τρίτη έκθεση που ετοιμάζει η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών για να αξιολογήσει το κατά πόσον υπάρχει διαφάνεια στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και ε, πρέπει να πω ότι εγώ ως εισηγήτρια και ως ευρωβουλευτής θεωρώ ότι η διαφάνεια είναι το κλειδί για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων πολιτών προς τα ευρωπαϊκά όργανα. Δυστυχώς βέβαια πρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η διαφάνεια μάλλον δεν έχει εγγραφεί ακόμα στο DNA μας. Ε, χρειαζόμαστε ε, και άλλο χρόνο διότι έχουμε πολύ περιττή μυστικοπάθεια. 85 τροπολογίες υπευλήθησαν, δεν θα σας τις αναφέρω μία προς μία. Φεύγω η κυρία Κοράτσα Μπίλ κρίμα, διότι ήταν μία από τις συντάκτρες των τροπολογιών. Οι άλλοι λείπουν ούτως ή άλλως, αλλά εγώ θα σας τα πω. Η κυρία Σόμερ υπέβαλε αρκετέ τροπολογίε. Φοβάμαι ότι αυτέ δεν θα μπορέσω να τι υποστηρίξω, διότι όλε προσπαθούν να μειώσουν την πρόσβαση στα έγγραφα και τη διαφάνεια. Θα μπορέσω να υποστηρίξω πολλές από τις τροπολογίες που υπέβαλε η κυρία Κοράτσα και η κυρία Μακοβάη, για παράδειγμα την έκκληση που κάνουν για να είναι διαθέσιμα έγγραφα στις ιστοσελίδες των θεσμικών οργάνων. Νομίζω ότι αυτό ε, θα μειώσει και τον αριθμό των ετοιμάτων που απευθύνονται προς τα όργανα για δημοσιοποίηση εγγράφων. Επίσης υποστηρίζω τι τροπολογίε του κυρίου Μόλτερ, ο οποίος μιλάει στο τηλέφωνο βέβαια τώρα. που κάνει έκκληση για μεγαλύτερη διαφάνεια σε ομάδες επιτροπολογίας και μια τροπολογία του κυρίου De Jong για την ε, δημοσίευση των πρακτικών των συνεδριάσεων των ομάδων Εργασία του Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων και των προτάσεων των κρατών μελών και τα ονόματα του μετά από την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού ε, δικαστηρίου για την ε, ε, υπόθεση για την πρόσβαση στις πληροφορίες και μπορώ να στηρίξω και τις τροπολογίες της κυρίας Αργεντίνη που ζητά από τα όλα θεσμικά όργανα να εφαρμόσουν τον κανονισμό για τη διαφάνεια κατά τρόπον ώστε να είναι συμβατά με την σύμβαση του Άρχους για περιβαλλοντικά ζητήματα και για τα I think those are my main remarks. Και για τα ανθρώπινα δικαιώματα νομίζω ότι αυτές είναι οι βασικές παρατηρήσεις που είχα να κάνω στους ελάχιστους που είναι εδώ στην αίθουσα. Η ψηφοφορία κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει στην Επιτροπή μας όχι στις 12 γιατί θα λείπω. Θα βρούμε μια άλλη μερομηνία, μάλλον στις 20 του μηνός και μετά θα προσπαθήσουμε να περάσει από την Ολομέλεια του Μαρτίου. Είναι κανείς εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριο Κρέγκερ θέλει να σχολιάσει, δεν είναι εδώ ο κύριο Κρέγκερ για να σχολιάσει. Αν δεν θέλει κάποιο άλλο το λόγο, όχι. Ωραία. Πιο σύντομο σημείο στην μερίσια διάταξη, μάλλον δεν ξαναείχαμε. Έχουμε μια ώρα μπροστά μας για το επόμενο σημείο. Και πάλι λοιπόν, για πέμπτη φορά σήμερα, διακόπτουμε μέχρι τις 4. Mm. Από ό,τι μου λένε, η κυρία Λεμπάη θα είναι εδώ στις 4, επομένως θα ήθελα να σας ζητήσω να έρθετε στις 4.